Ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Σας δίνω τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εψήφισαν 718. Άκυρες ψήφοι 35. Έγκυρες ψήφοι 683, 683 ψηφοδελτία γύρω. Η απόλυτη πλειοψηφία ως εκ τούτου ορίζεται, η απαραίτητη δηλαδή για την εκλογή σε πρώτο γύρο, στους, στις 342 ψήφους. Για την κυρία Φορέντσε ψήφισαν 50. Κυρία Λάμπερτς πήρε 56 ψήφους. Ο κύριος Πιτέλα 183. Ο κύριος Ρέμπιγκε

και ουδεμία υποψήφιος υποψήφια δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, θα περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θεωρώ πως παραμένουν ενισχύ οι υποψηφιότητες όπως είχαν ανακοινωθεί για τον πρώτο γύρο. Φορέντσα, Λάμπερτ, Πιτέλα, Ρέμπιγκα, Στέβενς, Ταγιάννη παραμένουν οι υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου. Μήπως θέλει κάποιος από τους α, συναδέλφους, των οποίων τα ονόματα εκφώνησα, να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Das ist nicht Όχι. Για το δεύτερο γύρο, λοιπόν, διατηρούνται όλες οι υποψηφιότητες δυνάμει του κανονισμού είναι δυνατό να κατατεθεί πριν από κάθε νέο γύρο νέα υποψηφιότητα. Υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να καταθέσει την υποψηφιότητά του για τον δεύτερο γύρο. Πρόεδρος, Θα ήμουν ε, ευγνώμων εάν για αυτή την τόσο σοβαρή διαδικασία που διοργανώνουμε δείχνατε και την ελάχιστη σοβαρότητα. Η προθεσμία λοιπόν για την ε, υποψηφιότητα για την κατάθεση υποψηφίων για τον δεύτερο γύρο ε, είναι μέχρι τις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στον προεδρεύοντα και μπορούν να κατατεθούν στον αναπληρωτή γενικό γραμματέα στο 00101. Είναι το γραφείο της Προεδρίας. Διακόπτουμε λοιπόν τώρα τη συνεδρίαση και ε, θα ήθελα να επανέλθετε στη μία η ώρα το μεσημέρι. Μία λοιπόν.